Ε, από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές την ενημέρωση για την εκλογή του κυρίου Κλίντς ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς αντικατάσταση του κυρίου Μικαέλ Τόιρερ από την 6η Νοεμβρίου 2015. Επίσης ε, ανακοίνωση εκλογής της κυρίας Νάτζια Χίρς Νάντζια Χίρς και Μάρτιν Σίρντεβαν όπως και Γιώργ Μόιτεν προς αντικατάσταση του Γκραφ Λάμστορφ, του Φάμπιο Ντεμάζη και της Φον Στόρτς από την 8η Νοεμβρίου του 2017. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους νέους συναδέλφους και να υπογραμμίσω ότι θα αναλάβουν τις θέσεις τους στο Κοινοβούλιο και θα συμμετέχουν σε όλα τα όργανα σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας.